Καλησπέρα σας. Ως Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, θα ήθελα να καλωσορίσω τα μέλη μας. Να καλωσορίσω θερμά την κυρία Λάρα, Υπουργό Εξωτερικών και, και Διεθνούς τη της Δημοκρατίας της Ονδούρας. Επίσης να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των διπλωματικών αποστολών τον κύριο Μαντρίτ, πρέσβη της Ονδούρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να καλωσορίσω επίσης τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Νταλαριτσία, προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και την Καραϊβική της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Η διαρμηνία θα παρέχεται στην στα αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, γαλλικά και πορτογαλικά και παθητικά στα ιταλικά. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω τα μέλη ότι η συνάντηση μεταδίδεται ζωντανά στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης σας έχει διανεμηθεί στα ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρηθεί ότι η ημερήσια διάταξη έχει εγκριθεί. Επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη ότι το Παρλασέν με την ευκαιρία της 60ης επαιτίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε δήλωση στις 17 Μαΐου του 2017 στην πόλη της Γουατεμάλας. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης στο φάκελο που σας έχει διανεμηθεί. Και στο σημείο αυτό καλωσορίζω την κυρία Αποέρο Λάρα, Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνού Συνεργασία τη Δημοκρατία τη και την ευχαριστώ για την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει μαζί τη. Κύριε Υπουργέ, Όπω γνωρίζετε, η αντιπροσωπεία μα έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα σα. Επισκεφτήκαμε, όπω θα θυμάστε, την Ονδούρα από τι 18 έω τι 20 Φεβρουαρίου του 2015 και κατά τη διάρκεια αυτή τη επίσκεψη η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία τη Ονδούρα, τον κύριο Χερνάντε, με εκπροσώπους της κυβέρνησης, του Κογκρέσου, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η αντιπροσωπεία ασχολήθηκε με μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων από οικονομικές και κοινωνικές πτυχές μέχρι την κοινωνική και νομική κατάσταση και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σας. Η επίσκεψη, αν και σύντομης διάρκειας, προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία στα μέλη της αντιπροσωπείας να εξοικειωθούν με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και να αξιολογήσει την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχαμε επίση την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την επιτυχή συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ονδούρα από πρώτο χέρι, όταν επισκεφθήκαμε δύο έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ένα για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών και το άλλο για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση στι λιγότερο αναπτυγμένε περιοχέ τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε επίση αποστολή παρατηρητών εκλογών για τι γενικέ εκλογέ τη 24η Νοεμβρίου του 2013 με την κυρία Λούνατσεκ, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως επικεφαλή παρατηρητή. Στα τέλη του 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε εκστρατεία παρακολούθηση των εκλογών στην Ονδούρα, με επικεφαλή επίση την κυρία Λούνατσεκ, για να διπιστώσει σε ποιο βαθμό οι συστάσει τη αποστολή παρατήρησης λήφθηκαν υπόψη. Μέσω τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρική Αμερική, η οποία κυρώθηκε την 1η Εβδόμου του 2013 στη χώρα σα. Οι σχέσει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ονδούρα, καθώ και με όλε τι άλλε χώρε τη Κεντρική Αμερική, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Σε όλε τι επισκέψει μου στην Κεντρική Αμερική, άκουσα την επιθυμία των χωρών για γρήγορη επικύρωση τη συμφωνία και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια προσωπικά έκανα ό,τι μπορούσα για να πείσω τα κοινοβούλια στα κράτη τη Ευρωπαϊκή μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνουν τη διαδικασία επικύρωση. Μέχρι και σήμερα, 21 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επικυρώσει συμφωνία, με τελευταία τη Λιθουανία, και προσδοκώ ότι τα υπόλοιπα κοινοβούλια θα ακολουθήσουν σύντομα. Ένα τομέα που απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα όπω και σε άλλε χώρε τη περιοχή. Η δολοφονία τη Μπέρτα Κασέρε στι 2 Μαρτίου του 2016 μα σώκαρε και ειλικρινά λυπούμαστε για το γεγονό ότι οι υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα δεν έχουν προσαχθεί ακόμα στη δικαιοσύνη. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τη σημερινή ευκαιρία ώστε να καλέσω εκ μέρους της αντιπροσωπείας τη σημερινή, την κυβέρνηση της Ονδούρας να κάνει ό,τι είναι δυνατόν εντείνοντας τις προσπάθειές της ώστε οι δράστες αυτής της δολοφονίας αλλά και παρόμοιων δολοφονιών κατά άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην μείνουν ατιμόρυτοι και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα να προστατευτούν από τέτοιες επιθέσεις στο μέλλον. Και εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε Σοφία Σακοράφα. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, πρέσβεις των χωρών της Κεντρικής Αμερικής και Λατινικής Αμερικής που βρίσκεστε εδώ, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των ε, πολιτών. Κυρίες και κύριοι, πολλοί από εσά επισκεφτήκατε τον Φεβρουάριο του 2015 την Ονδούρα. Η πρόεδρος, η κυρία Σακοράφα, που μόλις είχε αναλάβει την προεδρία της ΔΕΚΑΜ, ήρθε και ήταν πολύ σημαντικό που βρεθήκατε εκτεθειμένοι προσωπικά ο καθένας από εσά στα γεγονότα και στην πραγματικότητα της χώρας μου. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχτήκαμε εκεί και είχατε την ευκαιρία να ανταλλάξετε απόψεις με διάφορους παράγοντες της χώρας όσοι θέλαν να βρεθούν μαζί σας υπό τον Πρόεδρό μας Νολενάντες, Κοινωνία των Πολιτών και άλλοι. Από τότε βέβαια, από την επίσκεψη εκείνη μέχρι σήμερα, ο κόσμος βέβαια έχει εξελιχθεί κατά πολύ, έχει αλλάξει με τεράστια βήματα τα στρατηγική σημασίας προβλήματα οξύνονται, η τρομοκρατία έχει εξαπλωθεί με μεγάλη αγριότητα, το πανόραμα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι ένα πανόραμα χωρών και ομάδων χωρών που συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες και αρχές και εμείς πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι για να υποστηρίξουμε ένα δίκαιο μια δίκαια διεθνή τάξη που να, βασίζεται στα θεμελιώδη δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και την ακαιρεότητα των χωρών. Η Ονδούρα λοιπόν και η Κεντρική Αμερική είμαστε φίλοι, εταίροι, σύμμαχοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε από παλιά και από το 2014 με την ε, Συμφωνία Σύνδεσης που υπεγράφει στην Τεγουθικάλπα που είναι πρωτεύουσα της Ονδούρα προωθήσαμε ακόμα περισσότερο αυτή τη σχέση. Και είναι μια καλή στιγμή να επιταχύνουμε τώρα τη διαδικασία κύρωση της συμφωνίας αυτής σύνδεσης από τις χώρες μέλη εκείνες που δεν την έχουν ακόμα κυρώσει, όπως είπε και η Πρόεδρος. Σε αυτά τα δύο χρόνια επίσης η διεθνής κοινότητα επανεκατεύθυνε την στρατηγική της ανάπτυξη, οθετώντας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και προχωρώντας στους στόχους ανάπτυξης με μηχανισμούς καινοτόμους, πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και επίσης είχαμε και την εμβληματική COP21, τη συνεδρίαση αυτή στο Παρίσι και αυτό είναι ένα μόνο βήμα μπροστά που κάναμε αυτά τα δύο χρόνια. Πρόεδρε Σακοράφα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να οργανώσετε αυτή την έκτακτη συνάντηση ε, κατά την οποία θέλω να αποφεληθώ για να σας ενημερώσω για την κατάσταση στη χώρα μου, στην αγαπημένη Μονδούρα. Θα ήθελα να μιλήσω μαζί σας για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί επίσης στην ολοκλήρωση των χωρών της Κεντρικής Αμερικής και να σας ενημερώσω επίσης και για τις προοπτικές ανάπτυξης που έχουμε εμείς και για τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως λοιπόν έχουν προχωρήσει τα πράγματα στη διεθνή σκηνή, το ίδιο έχει συμβεί και στην ίδια τη χώρα, στην Ονδούρα, η οποία έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί. Είχαμε μια σημαντική πρόοδο όσον αφορά την κατάσταση λοιπόν στην Ονδούρα. Η πολιτική σταθερότητα πρώτα απ' όλα συνοδεύτηκε από ελπιδοφόρα οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε επίσης κοινωνικά επιτεύγματα στην υγεία, στην εκπαίδευση. Σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών. Δίνουμε περισσότερη προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο διάλογο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών. Επιτρέψτε μου τώρα, κάπω σύντομα, να αναφερθώ και σε κάποιου άλλους παράγοντε που είναι πολύ σημαντικοί στόχοι για μας. Πρώτα απ' όλα, στον πολιτικό τομέα. Πέντε μήνες πριν από τις γενικές εκλογές βρισκόμαστε για να εκλέξουμε πρόεδρο, βουλευτές και δημάρχους. Οι, προ... οι προκαταρτικές εκλογές κάθε κόμματος έγιναν τον Απρίλιο και η προετοιμασία των εκλογών ε, στην Ονδούρα από το 2009 έχει οδηγήσει σε νέες συμμαχίες που δεν είναι συνήθεις, ε, που είναι, δεν ήταν συνήθεις αλλά είναι συνήθεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας όμως είναι καινοτομία. Ε, ήδη έχουν ε, σχηματιστεί τρεις ε, πολιτικές δυνάμεις όσον αφορά την, την εκλογική αναμέτρηση και επικρατεί μεγάλος πολιτικός αναβρασμός. Ελπίζουμε ότι όπως και στις περασμένες γενικές μας εκλογές, θα στείλετε μια αναποστολή παρατήρησης των εκλογών για να παρακολουθήσει αυτή τη νέα εκλογική αναμέτρηση που είναι τόσο σημαντική για τον λαό της Ονδούρας, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής Αμερικής. Τώρα θέλω να έρθω στην οικονομία και την κοινωνική ανάπτυξη. Σήμερα η Ονδούρα έχει ενσωματώσει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στο δικό της σχεδιασμό εθνικό ανάπτυξης. Στην καθημερινότητα λοιπόν τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Είναι προσανατολισμός των δικών μας προτεραιοτήτων για να απαλείψουμε τη φτώχεια, για να μειώσουμε τις ανισότητες και να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Η δράση της κυβέρνησης της Ονδούρας βασίζεται στη δημιουργία ευκαιριών που επιτρέπουν την κινητικότητα και την κοινωνική συνοχή και αυτό μέσα από τη δημιουργία απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη με τη συμμετοχή όλων που να είναι και βιώσιμη. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ένα από τα στηρίγματα που έχουμε στο πρόγραμμα οικονομική μας ανάπτυξης που είναι το πρόγραμμα Οντούρα 2020 και βασίζεται στον τουρισμό, την υφαντουργία, την γεωργία, την μεταποίηση, τη στέγαση, τη στήριξη στο εμπόριο και θέλουμε με τον τρόπο αυτό να αναπτύξουμε μια παραγωγική πλατφόρμα και να βελτιώσουμε την διαγωνιστικότητα της χώρας μας, καθιστώντας την σε ένα ελκυστικό υλικοτεχνικό κέντρο στην περιφέρεια. Φέτος, το 2017, δημιούργηκαν 47.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Είχαμε πάνω από 190 εκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις εξαιτίας του προγράμματος αυτός και εξαγωγές της τάξης των 570 εκατομμυρίων δολαρίων. Από την περιφερειακή οπτική γωνία λοιπόν η Ονδούρα εξακολουθεί να προσφέρει στην θεσμική, στο θεσμικό καθεστώς του συστήματος ολοκλήρωσης στην Κεντρική Αμερική, το ΣΥΚΑ, και αυτό μέσα από την Τελωνιακή Ένωση ανάμεσα στην Ονδούρα και την Γουατεμάλα, κάτι το οποίο μας επέτρεψε να πετύχουμε 80% ε, ελεύθερες ε, συναλλαγές και ένταξη των ε, τριών τελωνιακών σταθμών ελέγχου των μεθοριακών και με δασμούς κοινούς κατά το 98%. Έτσι καταφέρουμε να μειώσουμε το κόστος κατά 25%, μειώνονται οι δαπάνες αλλά και ο χρόνος που χρειάζεται για τον έλεγχο στους μεθοριακούς αυτούς σταθμούς ελέγχου. Δεν πρόκειται για κάτι απομονωμένο από την ε, διαδικασία οικονομικής ε, ολοκλήρωσης. Βασιζόμαστε σε οικονομίες που λειτουργούν σε διαφορετικούς χρόνους και βασιζόμαστε στη συμπληρωματικότητά τους, με στόχο βέβαια τελικά να υπάρξει εναρμόνιση στην εμπορική μεταχείριση σε ολόκληρη την περιοχή. Και τώρα θέλω να έρθω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αποτελεί βασικό άξονα της ε, κυβέρνησης Ενάντες Αλβαράδο που έχει να κάνει με την θεσμική ενίσχυση και τη διακυβέρνηση. Η οικοδόμηση μιας δημοκρατίας περνάει από την προστασία των βασικών ελευθεριών και των ελευθεριών των πολιτών στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου. Εμείς πετύχαμε πρόοδο για να ενισχύσουμε τους θεσμούς που έχουν σαν σκοπό να διαλύσουν την διαφθορά και την ατιμορρησία που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη με τη βοήθεια της αποστολής για τη στήριξη του αγώνα κατά της διαφθοράς, που ονομάζεται MASIC, που είναι η πρώτη αποστολή της οργάνωσης των Αμερικανικών Οκροτών για να καταπολεμηθεί η διαφθορά σε μια χώρα μέλος. Και έτσι ενισχύσαμε την δικαστική θεσμικότητα και εξετάζουμε και ερευνούμε περιπτώσεις διαφοράς στην χώρα μας επιβάλλοντας κυρώσεις. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στη λειτουργία και στην αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού είναι κάτι που απέτησε βέβαια από κοινού προσπάθεια μεταξύ της κυβέρνησης και της ε, αποστολής αυτής για την καταπολέμηση ε, της διαφθοράς. Και έτσι καταφέραμε να πετύχουμε μηχανισμούς επιλογής δικαστικών φορέων, για παράδειγμα, να έχουμε ένα σύστημα πιστοποίησης των καταγγελιών, να δημιουργήσουμε μια πολιτική ποινική δίωξη κάθε φορά που έχουμε διαφθορά. Να υπάρχει επίσης ένα κανονιστικό πλαίσιο έρευνας για τα παραπτώματα, όπως είναι ο παράνομος εμπλουτισμός, να φροντίσουμε να υπάρχει η, καθαρή πολιτική, να εφαρμοστεί αυτή η καθαρή πολιτική, σαν τα καθαρά χέρια, και να δημιουργήσουμε, ε, να φροντίσουμε για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων. Αλλά πήραμε και άλλες πρωτοβουλίες, όπως την απόδοση λογαριασμών. Επίσης, έχουμε κάνει πρόοδο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε δημιουργήσει ένα θεσμικό δίκτυο προκειμένου να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και αυτών που τα υποστηρίζουν. Το άνοιγμα της κυβέρνησης λοιπόν επέτρεψε μια πολύ σημαντική παρουσία διεθνών οργανισμών. Πολλές φορές μας επισκέφθηκαν εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σαφές από όλα αυτά ότι έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να διασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών και να υποστηρίξουμε μια δημοκρατική ζωή. Βέβαια βασιζόμαστε γι' αυτό σε μία υπογραμματεία ειδική για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είμαστε στη διαδικασία να την κάνουμε γραμματεία από υπογραμματεία που είναι. Οπότε θα έχει δικό της προϋπολογισμό ήδη από το 2018. Έχουμε επίσης δημιουργήσει και γραφείο τη ΥΠΑ τη Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο ζήτησε η κυβέρνηση της Ονδούρα. Έχει υπάρξει δηλαδή πλήρες άνοιγμα για να έχουμε επισκέψεις από διεθνείς οργανισμούς και διαμερικανικούς και έχουμε λογοδοτήσει σε διεθνή φόρα. Η κυβέρνηση και η κοινωνία των πολιτών έχουν δημιουργήσει διάλογο για την εμπορία των ανθρώπων, για την προστασία των εκτοπιζομένων, για όσους είναι θύματα βίας, για όλους τους ευάλωτους, για όλες ευάλωτες ομάδες. Και για το 2016 έχει αποφασιστεί προϋπολογισμός 10 εκατομμυρίων λέμπαρες για να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα Τη νομοθεσία για την προστασία όσων ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφου κλπ. Και βέβαια είναι πολύ σημαντική σε όλα αυτά η συνεργασία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη σε αυτήν μπορέσαμε να προχωρήσουμε στους στόχους μας τους αναπτυξιακούς. Η συνεργασία με την Ονδούρα είναι μια καλή επένδυση. Η Ονδούρα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος, όπως φαίνεται και από το επιτυχές πρόγραμμα που έχουμε Κορεδόρ Σέκο και από την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επισητιστικής Ασφάλειας και Διατροφής. Έχουμε βοηθήσει 50.000 οικογένειες με μία πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν και άλλοι εταίροι για την ανάπτυξη και αυτό εξαιτίας των θετικών αποτελεσμάτων που είχαμε. Επίσης συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής μας υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης. Βάσει τα λόγια του Καουσίκ Μπάσου, που είναι οικονομολόγος και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, η απασχόληση είναι και η καλύτερη προστασία κατά της φτώχειας και της ευάλωτης θέσης. Και είναι κάτι που αναγνωρίζω και αναγνωρίζω τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κυβέρνησή μου, προκειμένου να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν οι κατάλληλε προϋποθέσεις. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι τα επιτεύγματα αυτά οφείλονται και στο σεβασμό των αρχών για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο φαίνεται σε καθημερινή βάση από τις σχέσεις της με την κυβέρνησή μας και φαίνεται και από τις εθνικές μας προτεραιότητες και από την συνέχεια που θέλουμε να δώσουμε στις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Και ως ε, τελικό σχόλιο θέλω να πω ότι σε θεσμικό επίπεδο σίγουρα Είχαμε στενές σχέσεις, πλούσιες, με περιεχόμενο και σημαντικές, με αποτελέσματα. Αλλά είναι οι προσωπικές σχέσεις που έχουμε σήμερα μεταξύ μας που είναι αναντικατάστατες. Θεωρώ ότι η δυναμική αυτή των προσωπικών σχέσεων και η δυνατότητα δράσης και αντίδρασης είναι αυτό που προσφέρει τη σωστή δόση αμεσότητας και πλουτίζουν το διάλογό μας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το διάλογο αυτό. Μακάρι να γίνει αυτό και πάλι στην Οδούρα, όπου μεγάλη χαρά θα σας υποδεχόμασταν ξανά στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε. Και πριν περάσω στους συναδέλφους για ερωτήσεις ή για σχόλια, να ρωτήσω την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αν θέλει να κάνει κάποια μικρά σχόλια ή τοποθέτηση. Κυρία Ανταλήρη Ευχαριστώ. Δεν έχω διερμηνία προς τα γαλλικά, αλλά μπορώ να μιλήσω γαλλικά από ό,τι έχω καταλάβει και νομίζω ότι θα καταλάβει ο υπουργό τι έχω να πω. Άκουσα στα αγγλικά, δεν είμαι σίγουρη ότι τα έχω ακούσει όλα. μου, πριν τοποθετηθείτε, πριν ερωτήσετε, θα πρέπει να τοποθετηθεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο Να εκφράσουμε τη χαρά μας για την ε, επίσκεψη της Υπουργού της Βρυξέλλες. Ε, με μεγάλη χαρά διοργανώσαμε την ε, συμμετοχή της Υπουργού στις Ευρωπαϊκές ημέρες Ανάπτυξης, όπου μπορέσαμε να έχουμε επικοινωνία μέσω ίντερνετ με την Ονδούρα με διάφορους δικαιούχους των project μας. Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ονδούρα είναι πολύ ανοιχτές, ειλικρινείς και θερμές. Και Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι προσκληθήκαμε για να στείλουμε αντιπροσωπεία παρατήρησης των εκλογών για τις επερχόμενες εκλογές. Ήδη έχουμε στείλει μία επιτροπή αναγνωριστικού τύπου που θα προετοιμάσει και το κείμενο επί το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για την αποστολή μιας ομάδας και ελπίζουμε πως θα θετικά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ πρόσωπε και τώρα τον λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Κυρία Ντορνάντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η φτώχεια πλήττει περίπου το 65% των οικοκυριών στην Ονδούρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ε, στην ύπεθρο σημαντικό. Πολλοί παράγοντες, όπως ε, είπατε, εξηγούν τον παράγοντα αυτό, επισφαλής εργασία, ε, οι δημόσιες υπηρεσίες, η ανασφάλεια κλπ. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ε, ποιες είναι οι πολιτικές που ασκούνται από την κυβέρνησή σας για να δράσετε αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες που οδηγούν στο φαινόμενο. Πολλά σκάνδαλα διαφθοράς δυστυχώς αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας της Ονδούρας έναντι των εκπροσώπων της κυβερνήσεως. Μετά, σύμφωνα με Transparency International, η αντίληψη που έχει ο πληθυσμό όσον αφορά τη διαφθορά έχει χειροτερέψει ε, κατά τη διάρκεια του 2000. Εδώ και δύο χρόνια βελτιώθηκε ε, και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Θα ήθελα να γνωρίζω με ποιους τρόπους θέλετε να καταπολεμήσετε τη διαφθορά. Επίσης, ε, να επιστήσω την προσοχή σας επί της αλλαγής του κλίματος. Εκεί η Κεντρική Αμερική ήδη υποφέρει από τις συνέπειες αυτές όπως είναι η ξηρασία και όπως είναι η ανύψωση του πιπέδου της θάλασσας. Η Γαλλία ανήκει σε αυτούς που συμφώνησαν στη, ε, υπέρ του συμφωνία του Παρισιού το 2015 ε, για το κλίμα. Μετά την απόσυση των ΗΠΑ από τη συμφωνία, κατά την άποψή σας, ποιο είναι το μέλλον των διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο για το κλίμα. Τέλος, με ενημέρωσαν για διάφορες ε, πιέσεις των δυτικών επί της Ονδούρας, ώστε η χώρα σας να υιοθετήσει κάποια ε, κάποια προσέγγιση, να εθετείς κάποια μέτρα για τις ε, εταιρείε. Είναι, αυτές οι πιέσεις είναι νομίμες. Η Ευρώπη και η Ονδούρα δεν έχουν τίποτα άλλο να μοιραστούν παρά αυτού του είδους θεωρίες. Ε, και το θέμα των φίλων χρειάζεται περισσότερη συνεργασία στο θέμα του πολιτισμού γενικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Η κυρία Αντιπρόεδρος για τη δική της ερώτηση, η κυρία Τσίντσι. Θα μιλήσω Ιταλικά, διότι από ό,τι κατάλαβα υπάρχει στα παθητικά. Θα μιλήσω Ιταλικά. Ευχαριστώ την Προέδρο, την κυρία Σακοράφα, για αυτή την συνάντηση και θα θέλω να χαιρετήσω την Υπουργό Εξωτερικών και να ευχαριστήσω για την παρουσία της εδώ, στη δική μας αντιπροσωπεία. Και θα ήθελα επίση ε, να την ευχαριστήσω για την παρουσίαση που έκανε για την πολιτική δραστηριότητα που γίνεται και τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει σε διάφορου τομεί η χώρα. Το Φεβρουάριο του 2015 είχα συμμετάσχει στην αποστολή ε, και είχα ήδη την ευκαιρία να εξακριβώσω τις προσπάθειες που καταβάλλονται στη χώρα, ούτως ώστε να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει ανάπτυξη. Ε, και συνάντησα διάφορες ενώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπόρεσα επίσης να συναντήσω νέους που ανήκουν σε διάφορους ε, οργανώσεις, σήμερα οργάνωση για την προστασία του περιβάλλοντος, που θεώρησα ότι ε, ήταν πολύ μαχητική στην προσπάθεια που κατέβαλαν. Και πήγαμε και επισκεφθήκαμε μια ένωση για την υπεράσπιση των γυναικών που ήταν αθήματα της βίας ήταν πάρα πολύ σημαντικέ στιγμέ που μα έδειξαν πόσε προσπάθειε καταβάλλονται στη χώρα σα. Εσεί το επιβεβαιώσατε αυτό, ενίσχυση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ενίσχυση των θεσμών, ε, οι προσπάθειε που καταβάλλονται για την καταπολέμηση τη διαφθοράς. Οι προσπάθειε για να επικρατήσει η διαφάνεια όσον αφορά τι δραστηριότητε τη κυβερνήσεω και τη διοίκηση. Σίγουρα αναμφισβήτητα αυτέ είναι πτυχέ σημαντικότατε Και χάρηκα που άκουσα και αυτό επιβεβαιώθηκε ότι ζητήθηκε μία αποστολή παρατήρηση όσον αφορά τις επικείμενες ε, ε, εκλογές. Πιστεύω ότι και αυτή είναι μία στιγμή πλήρους συνεργασίας μεταξύ της χώρας σας ε, και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η συνεισφορά που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα όμως ή δυνατόν αν επιτρέπετε να σας κάνω μία ερώτηση που αφορά μία πτυχή που στην αντιπροσωπεία το γνωρίζουν οι συνάδελφοι και που με ενδιαφέρει πολλά. Όσον αφορά τους ανήλικους, πιστεύω ότι η επένδυση στα παιδιά, επένδυση στους ανήλικους, που δυστυχώς είναι τα πιο άμεσα θύματα, τα πιο εύθραστα θύματα όσον αφορά τη φτώχεια, όσον αφορά τη βία, όσον αφορά το κίνδυνο να καταλήξουν στα χέρια ε, του οργανωμένου εγκλήματος που τα εκμεταλλεύονται για διάπραξη εγκλημάτων και δικημάτων και ο κίνδυνος των πιο μεγάλων παιδιών να μην βρούνε δουλειά. Στην Ονδούρα υπάρχει ένα φαινόμενο που δεν είναι μόνο φαινόμενο της χώρας σας, αλλά δυστυχώς ένα φαινόμενο διάχυτο των νέων ασυνόδευτων ανηλίκων, μάλλον ασυνόδευτων μεταναστών που εγκαταλείπουν τη χώρα για να προσπαθήσουν να βρουν δυνατότητα καλύτερης ζωής σε άλλες χώρες. Λοιπόν, ή θα σας ρωτήσω, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τα σχέδια εκπαιδεύσεως για τους ε, ανήλικους, για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος, οι κίνδυνοι αυτοί και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν περισσότερο οι ανήλικοι, διότι είναι και πιο ευάλωτα τα παιδιά, για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι μπορεί να αντιμετωπίσουν, θα πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση που στοχεύουν αποκλειστικά τους ανήλικους, όχι μόνο στο σχολείο, να του προσφέρουμε όμω και δυνατότητε, ούτω ώστε τα παιδιά να μπορούν να εκμεταλλευτούν τα ταλέντα τους, τις δεξιότητές τους και να μειωθεί ο κίνδυνος να μπλέξουν με το οργανωμένο έγκλημα και να καταλήξουν θύματα βιοπραγιών. Ε, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες συγκεκριμένε όσον αφορά αυτή την πτυχή. Η επένδυση στους ανήλικους, στους νέους, πιστεύω ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές ε, μορφές για να οδηγηθείτε στη σωστή ανάπτυξη της χώρας. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση έχω να σας κάνω και σας ευχαριστώ. Και εμείς κύριε Αντιπρόεδρε και το λόγο έχει ο κύριος Τέρι Καμπράς. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, που είστε σήμερα εδώ. Εσείς Είπατε κάποια πράγματα που πολύ με ενδιαφέρουν όσον αφορά κάποια από τα προβλήματα που έχετε είναι κοινά, κυρίως τα αρνητικά προβλήματα. Είναι προβλήματα τα οποία είναι κοινά σε άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Νότιας Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής. Υπάρχει όμως κάτι που με ενδιαφέρει εμένα όλος ιδιαίτερος και είναι αυτό στο οποίο εσείς αναφερθήκατε, ότι δηλαδή αποδίδεται μεγαλύτερη προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, όσον με αφορά δεν το αναλύσατε ιδιαίτερα ε, και δεν έχετε καταφέρει και πολλά πράγματα στην πράξη. Ελάχιστα θα έλεγα. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν αν έχετε τέτοια στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα κάποια στιγμή να έχω μια συγκριτική μελέτη, για παράδειγμα, για τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ονδούρα, για να δούμε τι έχει γίνει με την βία κατά των γυναικών, για παράδειγμα, ή με τις δολοφονίες τι γίνεται με την ατιμορρησία ή την αδικία. Και το λέω γιατί στις συγκριτικές μελέτες πάντοτε βλέπει κανείς την τάση που επικρατεί. Να δούμε αν είναι πραγματικά πολύ θετική ή αν βασίζεται μόνο όλη αυτή η προσπάθεια στην καλή θέληση, που είναι πολύ σημαντική βεβαίως, αλλά εδώ μιλάμε για πολιτικές και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε και πέρα από την καλή βούληση, την καλή θέληση. Το λέω γιατί η πρόεδρος ανέφερε την ε, αιματηρή δολοφονία της Μπέρτα Κάθερες που ήταν ε, τόσο εντυπωσιακή είναι μάλλον τόσο εντυπωσιακό που δεν έχει ακόμα βρεθεί ο ένοχος, δεν λύθηκε αυτή η υπόθεση και αυτό είναι ένα αρνητικό μήνυμα για το πώς προχωράει η δικαιοσύνη στην Ονδούρα, κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η τάση των τελευταίων ετών και επίσης τι μέτρα έχουν ληφθεί πρόσφατα στην Ονδούρα για να καταπολεμηθεί η διαφθορά, η ατιμορρησία και η βία και ταυτόχρονα να ευνοηθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν είναι νομικού τύπου, αν είναι κοινωνικού τύπου, αν είναι πολιτικού τύπου, αν είναι εκπαιδευτικού τύπου, τι είδους μέτρα έχουν δρομολογηθεί ή έχουν ειδηληφθεί, γιατί είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι η περάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι απλά ένα σήμα, ένα ε, σημεάκι που βάζουμε, όπως αυτά που βάζουμε πάνω στα κρουασάν, ή υπάρχει ή γίνεται, υπάρχει βελτίωση ή δεν υπάρχει. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα βέβαια μπορείτε να μου απαντήσετε αυτά που μπορείτε σήμερα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να δούμε ποιες είναι οι τάσεις, η εξέλιξη στην Ονδούρα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και περισσότερη αισιοδοξία τις εξελίξεις στη χώρα σας που τόσο αγαπάμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Κύριε Πρέσβη, επίσης, και όλους τους υπόλοιπους πρέσβεις και συνήθεις φίλους της αντιπροσωπείας μας για τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Σας χαιρετίζω εδώ. Και ιδιαίτερα χαιρετίζω αυτούς που δεν είναι εδώ συνηθισμένοι, τέσσερις από τη Γουατεμάλα προσκεκλημένοι που ήρθανε, ε, πρόεδροι, και διευθυντές από οργανώσεις. Καλώς ήρθατε όλοι στην συνάντηση αυτή. Και ελπίζω πολύ σύντομα να είσαστε εσείς εδώ στο βήμα και εσείς να μας διηγηθείτε τι συμβαίνει στις χώρες σας, ποιες είναι οι ανησυχίες σας κτλ. Κατόπιν τούτων. Και πάλι καλώς ήρθατε. Δεν πήγα εγώ στην Ονδούρα, δυστυχώς, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνω. Θεσμικά, νομίζω ότι με τη συμφωνία σύνδεσης έχουμε σχέσεις και όλοι το είπαν και η Πρόεδρος ότι όλοι τη θέλουμε και θέλουμε να κυρωθεί πλήρως από όλου. Δεν είναι εύκολο και έχει κρατήσει πολύ καιρό η διαδικασία, αλλά και εγώ πολύ θα ήθελα να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Τώρα διάφορα θέματα φίξατε και έχω... από διάφορες ερωτήσεις, αλλά υπάρχει κάτι που και εγώ θέλω να πω. Κάτι το οποίο πάντα συζητάμε είναι το θέμα της βίας και της διαφθοράς. Θα έλεγα ότι είναι μια υποχρέωση του κράτους να φροντίσει τα φαινόμενα αυτά να απαλληφθούν πλήρως από τη χώρα. Φαίνεται ότι υπάρχει μείωση των δολοφονιών, παραμένουν πολλές, αλλά οι στατιστικές τουλάχιστον αυτά λένε από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Ονδούρα, της Ονδούρα, ότι υπάρχει μείωση της τάξης 50%. Τόσο το καλύτερο. Θα έπρεπε να ήταν 100%. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό τουλάχιστον θέλουμε όλοι. Αυτό είπε και ο κύριος Στέρι Κουάμπρε. Θέλουμε λοιπόν να φέρει σε πέρας και την υποχρέωση αυτή η χώρα σας για πλήρη απάλληψη της διαφθοράς. Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο. Είχαμε ψήφισμα πριν από ένα χρόνο το πολύ, στο οποίο θέταμε διάφορα πολύ σοβαρά πράγματα. Πρέπει να λέμε τα θετικά όταν υπάρχουν και να επικρίνουμε τα αρνητικά όταν υπάρχουν. Λοιπόν, ε, απορρίπταμε με το ψήφισμα αυτό, τη δολοφονία κτλ. Και, και ζητούσαμε να υπάρξει έρευνα αλλά αυτό που δεν μας άρεσε είναι ότι δεν υπήρχε προστασία. Βέβαια θα απαντήσετε φαντάζομαι και σε αυτό γιατί σας γίνανε πολλές ερωτήσεις και θα απαντήσετε σε όλες. Πάντα εμείς θέλουμε προστασία και προστασία για άλλους. Ζούμε σε δημοκρατία, ελευθερία. Θέλουμε προστασία όλων των ανθρώπων. Τώρα πρέπει να υπάρξει πρόσκληση από εσά για να πάνε παρατηρητές για τις εκλογές σας. Οι εκλογές είναι αυτές που διασφαλίζουν την ελευθερία. Μιλήσατε επίσης για την ολοκλήρωση της Κεντρικής Αμερικής. και την πολιτική σταθερότητα. Είναι πολύ βασική. Πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα για να υπάρχει ανάπτυξη. Και μερικέ φορέ σε κάποιε περιοχέ του κόσμου δεν είμαστε συνηθισμένοι σε θεσμική σταθερότητα. Μιλάμε μόνο για πολιτική σταθερότητα και τελικά δεν καταφέρουμε να πετύχουμε την ανάπτυξη όπως θα τη θέλαμε. Θα ήθελα να αναπτύξω και άλλα ζητήματα για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή η σχέση αυτή και θα έπρεπε να βαγιωθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. να ξέρετε ότι έχετε την πλήρη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προχωρήσετε και να φέρετε σε πέρας το υψηφιστό καθήκον που είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να καταπολεμήσετε τη διαφθορά και τις δολοφονίες εννοείται και να βελτιωθούν και οι οικονομικοί σας δείκτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Τίποτα άλλο. Και τώρα πριν να ε, δώσω το λόγο στην κυρία Υπουργό για να απαντήσει στις ερωτήσεις, θα ήθελα, επειδή ακριβώς έχουμε πάρει ένα αίτημα από την εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών να παρέμβουν, να ρωτήσω τους συναδέλφους αν έχουν αντίρρηση να δώσουμε το λόγο. Συμφωνείτε κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Μάτο. Άρα λοιπόν... Εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Μάρτα Ιμπέρο, αλλά για πάρα πολύ λίγο, επειδή ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ περιορισμένος, στις 4 ακριβώς πρέπει να έχουμε τελειώσει. Δύο λεπτά εσείς και δύο λεπτά θα μιλήσει ο κύριος Μάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την αντιπροσωπεία. Ονομάζομαι Μάρτα Ιβέρα, εργάζομαι για τη ΣΥΦΚΑ και εδώ αντιπροσωπεύω εννέα διεθνείς ε, και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και δίκτυα που τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα. Υπάρχει πραγματική ανησυχία της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινή γνώμης και κοινωνία των πολιτών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα σας και γι' αυτό είναι και πολύ καλό που μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας ε, για τις σχετικές πληροφορίες ε, σας ευχαριστούμε με τη σειρά μας για τις πληροφορίες, για τα μέτρα που έχετε εφαρμόσει εκεί. Ε, δεν έχουμε ε, στοιχεία ωστόσο αρκετά για την μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα. Έχουν μεταρρυθμιστεί δύο είδους μεταρρυθμίσεις και εδώ οι διεθνείς οργανισμοί σχολίασαν το δύο αυτά είδη ποινικού κώδικα για την τρομοκρατία όπου οι τοβελινικές αυτών των κωδίκων ή άρθρων επιτρέπουν ε, μια περιοριστική ερμηνεία της εντολής των εκπροσώπων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει επίσης ομοφωνία από πλευράς της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, κοινωνίας των πολιτών αλλά και των θεσμών όσον αφορά την διερεύνηση της υπόθεσης της Περτά Κάθερες. Ε, ιδιαίτερα Χαιρόμαστε που στις έρευνες υπήρξαν κρατήσεις από, για μέλη της ίδιας της εταιρείας αλλά και του, από, από ε, τάξης των ε, ανώτατων στρατιωτικών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ε, ε, υπάρξει εξελίξεις. Ελπίζουμε ότι μέσα στο, σε αυτή την δικαστική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα καταφέρουμε, καθώς είναι έτοιμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μέσω μιας ενός ψηφίσματος, να μπορέσουν να βρεθούν και να συλληφθούν και οι ηθικοί αυτούργοι. Ευχαριστώ, Αλκάρι. Θέλω να αναφερθώ κι εγώ στην κατάσταση όσων υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Μισελ Φόρ και ο κ. Αρόσκο τον Αύγουστο του 2016, εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Συστήματο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κεντρική Αμερική, είπαν ότι η Ονδούρα ήταν μια από τι πιο επικίνδυνε χώρε όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε στοιχεία από το 2001 κάθε χρόνο έχουμε τουλάχιστον έναν που χάνει τη ζωή του εξαιτία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2015 όμως έχουμε στοιχεία που βλέπουμε ότι κάθε μήνα έχανε τη ζωή του κάποιος που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε και χαιρόμαστε που υπάρχει αυτό το σύστημα προστασίας τώρα των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων, αλλά έχει και πολλές ελλείψεις και δυναμίες. Δεν υπάρχει προσφυγή και εξαρτάται πολύ από την αστυνομία και όχι από άλλες δομές. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο μηχανισμός αυτός προστασίας. Κάτι άλλο που μας ανησυχεί επίσης και που συμβαίνει και σε άλλες χώρες της περιοχής είναι ε, το θέμα της θετικοποίησης. Η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να είναι στα χέρια της αστυνομίας, όχι των στρατιωτικών αρχών. Και στην Ονδούρα και σε άλλες χώρες πρέπει όλο και περισσότερο να είναι η ασφάλεια αυτή όντως στα χέρια των αστυνομικών και όχι των στρατιωτικών. Και τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δολοφονήθηκαν συνεργάζονταν με άλλους ακτιβιστές υπέρ του περιβάλλοντος, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη σύσταση των Ηνωμένων Εθνών για τους ε, πληθυσμούς τους αυτόχθονες που λέει ότι πρέπει να είναι ενημερωμένοι οι αυτόχθονες πληθυσμοί για το τι θα συμβεί με την γη στην οποία ζουν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, ολόκληρα Ένα διαδικαστικό, λέει ο κύριος Φυσικά, εδώ πέρα είμαστε σε δημοκρατία και όλοι μπορούν να πούν ό,τι θέλουν, αλλά εγώ δεν είπα ότι είμαι κατά του να πάρουν το λόγο οι εκπρόσωποι της κοινωνίας ε, των πολιτών, αλλά να μην έχουμε τέτοιες ε, εκπλήξεις. Εδώ είμαστε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε ευρωβουλευτές εδώ για ένα συγκεκριμένο θέμα. Και εντάξει, συμφωνώ να προσκαλούμε όποτε θέλει να έρχεται η κοινωνία των πολιτών εδώ και όποιο θέλει να παρακολουθεί. Αλλά λέω ότι δεν είναι σωστό να έχουμε τέτοιες εκπλήξεις. Τώρα δεν θα έχουμε χρόνο, έχουμε 8 λεπτά μόνο για να απαντήσει η Υπουργό. Η κοινωνία των πολιτών είναι τελευταία που παίρνει το λόγο. Δεν έχει νόημα, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα αυτό στο μέλλον να το διευθετήσουμε διαφορετικά. Ευχαριστώ για τους προβληματισμούς σας. Δεν τους συμμερίζομαι. Κύριε Μάτο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. τήρησα τη διαδικασία. Πήρα ένα αίτημα, είμαι υποχρεωμένο να το θέσω στο σώμα, το έθεσα, το αποδεχθήκατε. Το τι θα πει ο καθένα όταν λάβει το λόγο είναι δικό του πρόβλημα. Το θέμα είναι να μπορεί και να έχει το χρόνο να απαντήσει η κυρία Υπουργό. Νομίζω ότι έχει δέκα ολόκληρα λεπτά και μπορεί να απαντήσει. Δεν νομίζω ότι δικαιούμαι ω πρόεδρο να θυμώσω, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά οποιονδήποτε παίρνει το λόγο. Είτε είναι συνάδελφο, είτε είναι κάποιο ο οποίο έχει ζητήσει το λόγο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να είμαι κάθετη. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. de un compartir que ha querido ε, κοιτάξτε, είμαστε χώρε ε, φίλοι, αλλά η κοινωνία των πολιτών είναι παρούσα στην Ονδούρα παντού, σε διάφορα κυβερνητικά, κρατικά α, θεσμικά όργανα, ε, το πολιτικό, το δικαστικό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας και μάλιστα εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι είστε σήμερα, ότι είστε μάλλον παρόντες μονίμως στην Ονδούρα Δεν μπορώ παρά να σας, να ενημερώνω και να μπορούμε να μοιραστούμε και τις προσπάθειες που καταβάλουμε. Είμαστε μια μικρή χώρα. Η καλή θέληση δεν αρκεί όμως όπως είπατε κύριε Κάμπρας. Είμαι βεβαία ότι η καλή θέληση δεν αρκεί σε μια χώρα που έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες προκλήσεις όπως αυτές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς στην Ονδούρα ή σε οποιαδήποτε χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συζητήσουμε και θα ήταν ε, ε, ανόητο να πει κανεί ότι μόνο με την καλή θέληση μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Έχουμε καταλόγους με συγκεκριμένες δράσεις με τις οποίες έχουμε προβεί σε αυτήν την ε, αλλαγή. Μπορώ να, έχω κατάλογους, λοιπόν, μπορώ να σας τα αφήσω να δείτε και να αναλύσετε πραγματικά και να μπορέσουμε έτσι να ανταλλάξουμε απόψεις και με τους ε, πρέσβεις, σα ε, πρέσβεις των χωρών σας στην χώρα μου. Κοινό παρονομαστή για όλου είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα τη Μπέρτα Κάθερε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για εσά, αλλά και για μένα, που είμαι από την Ονδούρα και είμαι και γυναίκα και είναι απαράδεκτο να λέμε ότι στο τέλος της ε, διαδικασίας δεν είχαμε αποτελέσματα. Είναι απαράδεκτο. Οχτώ άνθρωποι φυλακίστηκαν στην ε, διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας. Είναι οι δράστες. Εμπιστεύομαι ε, απόλυτα το Σύνταγμα μας και τη συνταγματικότητα των όσων συμβαίνουν εκεί. Καμιά χώρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δικαιοσύνη μας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό που ο πρόεδρος ανέλαβε πρωτοβουλίες που ήδη τι ανέφερα, αλλά μπορώ και να τις επαναλάβω αν το επιθυμείτε, την ε, καθίδρυση του ΙΣΥΠΑ τη Αρμοστία ε, που σας ενημερώνει για τις πρόοδου αυτέ την ε, καθίδρυση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη Ατιμορρυσία, που είναι παρούσα σε όλες τις ακροηματικέ διαδικασίες ε, τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισπανίας που ήταν εκεί παρόντες ε, και στην ακροαματική διαδικασία για να ασχοληθούν με το θέμα των τεσσάρων αυτών κρατούμενων των οποίων η ακροματική διαδικασία έχει προβληθεί για την επόμενη εβδομάδα. Επιμένουμε ώστε να, βρεθεί, να βρεθούν οι ένοχοι. Εγώ πρώτη από όλου ενδιαφέρομαι στο να φτάσουμε στην επίλυση το, και να βρεθούν οι ηθικοί αυτούργοι. Όμως θα πρέπει να έχουμε το σωστό συνομιλητή ώστε να έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες για αυτές τις υποθέσεις ε, είναι η κυβέρνηση της Ονδούρα. Πολλές φορές ε, άλλες φωνές ακούγονται πιο δυνατά από τη δική μας και γι' αυτό και σήμερα είμαι εδώ ενώπιόν σας ώστε να επικρατήσει διαφάνεια για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε, να ακούσω τις ανησυχίες σας και πάνω απ' όλα έτσι ώστε μια χώρα και ένας εταίρος τα χώρες μέλη της Ένωσης και ένας ε, ε, εταίρος όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση των θεσμών ε, στην Ονδούρα. Νομίζω πως όσον αφορά τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα είμαστε στο σωστό δρόμο. Οι κόρες της κυρίας Κάθερες ε, βρήκαν ανοιχτέ τις πόρτες σε όλους τους θεσμούς όπου ε, ζήτησαν να βρίσκονται παρούσες, είναι παρούσες σε ακροματικές διαδικασίες της δίκης και Όποιο γνωρίζει σε ποια κατάσταση είναι η χώρα μου γνωρίζει πω έχει υπάρξει πρόοδο. Έχουν ακόμα πολλά να γίνουν, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν πρέπει να χάνουμε την εμπιστοσύνη μα. Δεν θυμάμαι τώρα αν έγινε κάποιο άλλο σχόλιο σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να αναφερθώ και στην ΣΥΦΡΕ, γιατί υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί όπως η Global Witness που ήρθαν στη χώρα μου και ε, τα νούμερα που δίνουν ε, ε, δίνουν ε, το 400% της πραγματικότητας στη χώρα μου. Ο συνομιλητής σας λοιπόν θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η κυβέρνηση της χώρας, η Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μόλις λάβαμε μάλιστα απόφαση να την τοποθετήσουμε σε υπουργικό επίπεδο και επίσης ε, συμμετέχουν ε, ε, αντιπροσωπείες μάλλον ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Επιτροπή αυτή. Και μάλιστα και εγώ είμαι πλήρες μέλος της Συμβουλίου Προστασίας των Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε ε, επίσης συμμετοχή του εις των Δημοσιογράφων, εκπροσώπους της κοινωνίας των ε, πολιτών, των αρμόδιων υπουργείων και άρα η αποφασιστικότητά μας είναι να προχωρήσει η χώρα μας. Και αυτό μόνο ο λαός μας μπορεί να το καταφέρει. Ε, τώρα θέλω να αναφερθώ στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Ήδη το ανέφερα προηγουμένως ότι ε, με δεδομένων αυτών των ε, υποθέσεων των εμβληματικών που αναφέρατε, υπήρξε ένα κίνημα στη χώρα μας που απέτησε μια μόνιμη αποστολή στη χώρα για να διερευνηθούν αυτές οι υποθέσεις διαφθοράς. Ε, επί τη βάση αυτού του αιτήματο, η κυβέρνηση της Ονδούρας ζήτησε τον προσανατολισμό και τη στήριξη του Οργανισμού των Αμερικανικών Κρατών που μάλιστα παρουσίασε μόλις τη δεύτερη του έκθεση όσον αφορά τις ε, ε, ε, διάφορα νομοθετήματα όπως ο νόμος για την καθαρή πολιτική στις επόμενες εκλογές μας ε, μάλιστα θα ολοκληρωθεί και θα εγκριθεί αυτή η νομοθεσία και είδαμε ότι πρόκειται για μια αποστολή στην ουσία ένα σώμα το οποίο στην ουσία στηρίζει το ανώτατο δικαστήριο, στηρίζει το Υπουργείο να ενισχύσει τις δυνατότητές του. Και γιατί το λέω αυτό. γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει εμείς οι ίδιοι να κάνουμε. Μπορεί να μα βοηθήσει στο να αναπτύξουμε δυνατότητες και μετά θα πρέπει αυτός ο εκάστοτε θεσμός που μας βοηθάει να αποσυρθεί από τη χώρα, αφήνοντας ε, τους κρατικού μηχανισμούς όμως ισχυρότερους. Αυτές είναι οι εκθέσεις λοιπόν που έχουν ε, ήδη ε, παρουσιαστεί στον Οργανισμό Αμερικών Κρατών. Πριν από ένα μήνα μόλις παρουσιάστηκε η τελευταία έκθεση όπου γίνεται και μία δήλωση ε, πολύ σοβαρή της κυβέρνησής μας για δέσμευση στις γραμμές που υπέβαλε αυτήν η αποστολή ε, τις οποίες δεσμεύεται να ακολουθήσει η κυβέρνηση της Ονδούρας. Τώρα, κλιματικές αλλαγές. Είμαστε μια από τις πιο ευάλωτες χώρες του κόσμου στις ε, κλιματικές αλλαγές. Η Ονδούρα είναι μια από τις 147 χώρες που έχουν ε, συνυπογράψει την, ε, και κυρώσει τη συμφωνία. Το κάναμε μάλιστα άμεσα γιατί πρόκειται για μια δέσμευση του Προέδρου μας η Ονδούρα επηρεάζεται όπως και άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής ε, σε αυτό που ονομάζεται ο ξηρός διάδρομος και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βοηθά ενεργά για την διατροφική ασφάλεια των οικογενειών που βρίσκονται και ζουν σε αυτή τη ζώνη και μάλιστα μέσα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ε, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και ελπίζουμε πως οι χώρες που ήδη έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης ε, ε, θα συνεχίσουν και αυτές και κάτι ακόμα το οποίο θέλω να θέσω και είναι στο μυαλό όλων μας είναι το θέμα της αρχής της ευθύνη. Εμείς ε, επηρεαζόμαστε από τις συνέπειες των ε, κλιματικών αλλαγών χωρίς να είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτές τις κλιματικές αλλαγές και μάλιστα έχουμε ε, συντάξει το σχέδιο ε, για το νερό, τα δάση και τα εδάφη είναι ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει διάφορες δράσεις για μεγάλα κομμάτια της χώρας και εθνικού τύπου δράσεις που εμπίπτουν μέσα στο πλαίσιο των διεθνών μας αυτών δεσμεύσεων. Ναι, και νομίζω πως δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά ότι ανέφερα αυτά που με ρωτήσατε. Και όπως είπα και στην αρχική μου εισήγηση, θα ήθελα να έρθετε να γνωρίσετε τη χώρα μου για να διαπιστώσετε τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει και το είπαμε και χτες στον ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στο πλαίσιο του European Development Days τις Ευρωπαϊκές ημέρες Ανάπτυξης όπου είδαμε, είχαμε τη μαρτυρία σχεδόν 30 συμπατριωτών μου που παρουσίασαν την εμπειρία τους και τα καλά αποτελέσματα από τα διάφορα προγράμματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, Ονδούρα που βοηθάει πραγματικά τη μεταμόρφωση τη χώρα μας και την οικοδόμηση της νέας Ονδούρας που όλοι επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι είναι ικανοποιημένοι από τις ε, απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις που σας θέσανε. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχετε πάρει απόφαση να προχωρήσει η χώρα και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μονάχα με τη συμμετοχή του λαού. Έχετε μπροστά σας μια πολύ σημαντική διαδικασία, δημοκρατική διαδικασία που είναι εκλογέ από καρδιάς. Προσωπικά σας εύχομαι, αλλά πιστεύω και οι συναδελφοί όλοι. Καλή επιτυχία σε αυτές τις εκλογές και στο επανειδήν. Ε, θα ήθελα, εδώ τελειώνει φυσικά η συζήτησή μα και θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη ότι η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση αντιπροσωπεία μα θα πραγματοποιηθεί την 5η στι 22 Ιουνίου του 2017 στι Βρυξέλλε. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και του μεταφραστέ και για την παράβαση που κάναμε και την υπέρβαση στον χρόνο.